colleagues. Συνάδελφοί μου, αν δεν απατώμε μπορούμε να αρχίσουμε. Τι να αρχίσουμε, τη συνεδρίασή μας. Στο σημείο 9 βρισκόμαστε. Καλωσορίζουμε εδώ τον Ιωνάθαν Χίλ δική μας συνεδρίαση ο Επίτροπος Χίλ έχει εμφανιστεί και το Φεβρουάριο για να παρουσιάσει την πράσινη βίβλο για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών. Είχαμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση και τότε, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεται για πλήρη ανταλλαγή για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του από τότε που ανέλαβε. Καλωσορίσατε κύριε Επίτροπε διαβάσαμε την πράσινη βίβλο με μεγάλη προσοχή. Είχαμε και μία πρώτη απάντηση ως ψήφισμα, με μορφή ψηφίσματος που θα εγκριθεί ελπίζουμε το Μάιο. Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τις επιπτώσεις της ε, νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με εισηγητή τον συντονιστή του ΕΛΚ κ. Μπάλς και θα θίξουμε και τα γενικότερα θέματα που θέτει η πράσινη βίβλος όπως πώς να εξισορροπήσουμε την σταθερότητα με την ανάπτυξη που είναι γενικότερο και ζωτικό θέμα. Ξέρω ότι και εσείς ενδιαφέρεστε και το προσέχετε ιδιαίτερος. Και θα προσεχθεί επίσης ιδιαίτερα τους επόμενες εβδομάδες και μήνες όταν θα συζητιέται, συζητούνται συγκεκριμένα πτυχές της πραγματοποίησης, υλοποίησης της Τραπεζικής Ένωσης. Υπάρχει και η έκθεση Γκουλάρ για το ρόλο της Κομισιόν στα διεθνή βήματα και αυτό ωραίο θέμα. γιατί ξέρουμε ότι σε εκείνο το επίπεδο γίνονται χρήσιμες συστάσεις πάντοτε. Και επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω δύο θέματα πριν σας δώσω το λόγο. Πρώτον, πρέπει να προχωρήσουμε επί όλων των προτάσεων που εκκρεμούν από την προηγούμενη θητεία μετά την επιτυχή διαπραγμάτευση του ΕΛΤΙΦ του ξεπλήματος προμήκου χρήματος πρέπει να προχωρήσουμε και για την οδηγία των πληρωμών ψηφίσαμε ήδη στην Επιτροπή τον Απρίλιο θα ψηφιστεί και στην Ολομέλεια. Ελπίζουμε να μας υποστηρίξετε όταν ζητήσουμε από το Συμβούλιο στεναρή δέσμευση για όλα αυτά τα θέματα που συνδέονται φυσικά με τη σταθερότητα. Εξάλλου η εικόνα θα ψηφίσει τώρα σε λίγο για θέματα διαφάνειας κλπ. Και την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε για την πρόταση benchmark και το ζωτικό θέμα της μεταρρύθμισης τραπεζικού τομέα. Υπολογίζουμε σε εσά λοιπόν και την Επιτροπή γενικότερα, την Κομισιόν, για να γίνουν όλα αυτά νόμος. Έπειτα είδαμε το πρωί, συζητήσαμε μάλλον το πρωί με την Κομισιόν και με το ΕΣΜΑ άλλα σημαντικότατα μέτρα και είναι φανερό ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μας. Ξέρω τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί, η Κομισιόν και οι υπηρεσίες της και εμείς που πρέπει να αντιμετωπίσουν τον τεράστιο φόρτο εργασίας. Το Κοινοβούλιο θα διαθέσει περισσότερους ανθρώπινους πόρους και για τις κατεξουσιοδότησης πράξεις, αν και δεν έχουμε και πάρα πολλούς. Το θεωρούμε πολιτική παρατεραιότητα και ελπίζουμε η εξαιρετική μέχρι τώρα συνεργασία μας να συνεχιστεί και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγή. Με μεγάλη χαρά έρχομαι ένα μήνα μετά την περασμένη μας συνεδρίαση για να συζητήσουμε την Πράσινη Βίβλο για την Ένωση Κέφαλαια Αγορών. Ε, θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και ε, θα αναφερθώ ενδεχομένω στα σχόλιά σα που ήταν πολύτιμα. Σήμερα χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να συζητήσουμε ευρύτερα όλο το φάσμα για να σας ενημερώσω για ορισμένε πρόσφατε εξελίξεις. Πριν το πράξω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα πολλά μέλη της Επιτροπής σας, με τα οποία είχα πολύ χρήσιμες και γόνιμες συζητήσεις από τον Νοέμβριο ε, ε, χαίρει πολύ ψηλής εκτίμησης η Επιτροπή σας. Ακούσαμε ε, ε, πόσα θέματα χειρίζεστε και κατάλαβα κι εγώ ο ίδιος για ποιο λόγο χαίρεται τέτοια εκτίμηση. Στην ακρόαση μου πέρυσι έθεσα πέντε τομείς προτεραιοτήτων, εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της τελευταίας πενταετίας, ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν, ε, εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής εφαρμογής διεθνών προτύπων και αρχών, ανάπτυξη της ε, Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών και επέκταση των ωφελιών ε, της εσωτερικής αγοράς πιο άμεσα στους πολίτες. Να σας αναφέρω λοιπόν τι κάνουμε σε αυτούς τους πέντε βασικούς τομείς. Πρώτον, για την εφαρμογή και πιο σημαντικό είναι η Τραπεζική Ένωση εδώ. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά και πρόοδο. Ο μηχανισμός SSM ανέλαβε 1η Νοεμβρίου την εποπτεία με ε, την ε, υποστήριξη της Επιτροπής σας. Ορίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρετικούς εκπροσώπους στον υποπτικό μηχανισμό. Αύριο συνεδριάζει για πρώτη φορά σε Ολομέλεια. Πριν από τα Χριστούγεννα ε, συμφωνήσαμε πόσα θα δώσουν τα κράτη-μέλη στο ενίο Ταμείο Εξηγένσης και ε, τώρα θα πρέπει η BRD να ε, μεταφερθεί και η διακυβερνητική συμφωνία να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη. Το είπα αυτό στην τελευταία συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω σήμερα ότι δεν θα χαλαρώσω την πίεσή μου. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ε, μέτρων επίπεδου 2, στα οποία μόλις αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, ξέρετε ότι είναι τεράστιο αυτό το έργο της προώθησης. Είναι πάνω από 400 αρμοδιότητες του ε, επίπεδου 1 και θα γίνουν 345 φέτος. Και σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες του επίπεδου 2 βεβαίως θα σεβαστούμε το πρώτο επίπεδο και θα πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή ανάμεσα ε, στη διαχείριση κινδύνου και την αναλογική αντιμετώπιση. Με τη συμμετοχή της ομάδας εμπειρογνωμών νομίζω το Κοινοβούλιο έχει από την αρχή ε, συμπεριληφθεί στην εκπόνηση κατεξουδότησων πράξεων και ε, οι τεχνικές προδιαγραφές επίπεδο προσχεδίου από τις εποπτικές αρχές ε, υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια στους συνομοθέτες. Έχουμε ε, μηνιαίο έλεγχο στα μέτρα του επίπεδου 2 και εγώ διμερείς συνεδριάσεις και επαφές με τους εισηγητές για να συζητήσω θέματα ενδιαφέροντος της κάθε Ελπίζω αυτές οι συνεργασίες να είναι χρήσιμες και να λειτουργούν καλώς. Τώρα, στο δεύτερο τομέα θα ήθελα σύντομα να σας ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε ε, με τα θέματα που εγώ κληρονόμησα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λαμασούρ και τον αντιπρόεδρο κύριο Σάλβα για τα LTIFs και το MIF, ε, το αντίστοιχο κανονισμό. Σε ό,τι αφορά τα LTIFs, ε, το αυτό που με ενδιαφέρει είναι πολύ γρήγορα να τεθούν σε ισχύ και φέτο ε, οι κανόνε του επίπεδου 2 για να έχουμε ασφάλεια δικαίου και να μπορούν οι επιχειρήσει να, να αρχίσουν να ε, πουλούν αυτά τα προϊόντα σε επενδυτέ και έτσι θα δημιουργηθούν δευτερογενείς ε, αγορές για έργα υποδομών ή για δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέλω γρήγορα να προχωρήσουμε. Όπως ξέρετε, σε τριμερή διάλογο συζητούνται διάφορες προτάσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την επικοδομητική της συμμετοχή στους πολιτικούς τριμερείς διαλόγου στην αναθεώρηση της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση για τις ασφάλειες. Ευχαριστώ τον κύριο Λάγκεν και την οδηγία για τις υπηρεσίε πληρωμών. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη. Γνωρίζω ότι οι συζητήσεις ήταν επικοδομητικέ και έχουν δώσει ένα ε, πλαίσιο κοινή ε, κατανόησης για τα θέματα και συμφωνίας που πρέπει να προωθηθούν. Θα συνεχίσουμε και σε επίπεδο πολιτικό και σε τεχνικό να βοηθούμε και θέλουμε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια υπό λετωνική προεδρία. Σε ό,τι αφορά ε, τα ταμεία χρηματαγορών. Ε, χαίρομαι ότι δεν ήταν εύκολο και θέλω να συγχαρώ την Ιναγκήλ για τη συμφωνία που επετέφθη στην Επιτροπή σας. Τώρα εναπόκειται στο Συμβούλιο να συμφωνήσει για μια γενική προσέγγιση. Ο δικός σας συμβιβασμό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντιμετωπίζει κάποιες από τις ανησυχίες ε, για τα MMF και τον κίνδυνο ε, μετάδοσης μεταξύ τραπεζών και των ταμείων χρηματαγορών. Χαίρομαι για την ε, απόφαση που πήρατε για τη ρευστότητα, για ε, τι ναι, απαιτήσει για τη διαφάνεια. Τώρα κοιτούμε ε, το κατόφλι για 20 μονάδες βάσης για τα ε, και τα SINAF. Γνωρίζω επίσης ότι συζητάτε αυτό το καιρό διάφορες εκθέσεις για την χρηματοδότηση του κυρίου Σόρου ε, τα benchmarks ε, της κυρία Πανόεν Χόισε, του κύριου Χιόκμαρκ, την έκθεση και την επαγγελματική σύνταξη του κύριου Χέις. Εκτός από αυτά τα σημαντικά θέματα θα πρέπει να παραμένουμε ε, σε επαγρύπνηση γιατί ενδεχομένως να αναδύονται νέοι κίνδυνοι και ρίσκα. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει προτάσεις για την ε, ανάκαμψη και, και εξυγίανση μη τραπεζικών ιδρυμάτων. Να σας πω τώρα δύο λόγια για την τρίτη προτεραιότητα, διεθνείς προδιαγραφές και αρχές διεθνή πρότυπα. Θα πρέπει να υπάρξει μια σταθερή και σωστή εφαρμογή αν θέλουμε να βοηθήσουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να αποφύγουμε την κανονιστική διατησία και να υπάρχει δυνατότητα άνθησης της διασυνοριακής χρηματοπιστωτικής δράσης. Έχουμε κανόνες για το κεφάλαιο και για τη ρευστότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ε, διστάζει να εφαρμόσει τα διεθνή πρότυπα με τρόπο που να έχει νόημα για την Ευρώπη και που να ανταποκρίνεται στο διαφορετικό τοπίο που έχει η Ευρώπη. Είμαστε πολύ ανοιχτοί απέναντι σε άλλες δικαιοδοσίες. Βεβαίω εφόσον υπάρχουν ίσοι κανόνες παιχνιδιού είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις αγορές μας για επιχειρήσεις από τις τρίτες χώρες. Και αυτό αντιστοίχω προβλέπεται. Οι υπηρεσίε μου εργάζονται με τι Ευρωπαϊκέ Εποπτικέ Αρχέ για να επιληφθούν των τεχνικών αξιολογήσεων που χρειάζονται για να ληφθούν αποφάσει για τρίτε χώρε. Και η αντιστοιχεία, η αμοιβαιότητα δεν είναι ε, γραμμή, ε, ε, γραμμή νομοθετική σύγκριση, αλλά έχει σημασία αναλογικότητα. Υπάρχουν διαφορέ από χώρα σε χώρα βεβαίω ανάλογα με το μέγεθο και την παγκόσμια παρουσία της. Τον περασμένο μήνα είμαι στι Ηνωμένε Πολιτείε και χαίρομαι που μπορώ να σα πω ότι στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στην αντίστοιχη ρύθμιση ε, Έχουμε περισσότερα που μα ενώνουν και λιγότερα που μα χωρίζουν με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Καμιά φορά όμω, ε, μέχρι τελευταία στιγμή αγωνιζόμαστε, όπως ήταν στη διαπραγμάτευση για το CFTC ε, για ε, συναλλαγές διασυνοριακές παραγόγων. Δεν χρειάζεται να έχουμε ακριβώς τους ίδιους κανόνες, αλλά θα βοηθούσε αν υπάρχει ένα στεναρό σύστημα συνεργασίας νωρίς στην ρυθμιστική διαργασία. Και έρχομαι τώρα στο TTIP που γνωρίζω συζητείτε κι εσείς αυτό τον καιρό με τον εισηγητή σας, τον κύριο Κόφοντ. Πιστεύω λοιπόν ότι η καλύτερη συνεργασία θα μας βοηθήσει να ε, ε, εγκαθιδρύσουμε τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Πολιτειών με διεθνείς κανόνες που θα τους εφαρμόζουμε με συνέπεια και στενή εποπτική συνεργασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να βασίζονται ο ένας στους κανόνες του άλλου εφόσον έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα θα μειωθεί το κόστος και οι τριβές που δυσκολεύουν τη ζωή για μια παγκόσμια δράση και ε, εμποδίζουν ε, τον κόσμο από τη συμμετοχή σε αυτό το σύστημα. Επίσης αυτό θα έχει και μεγαλύτερες εγγυήσεις για χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ε, συνεργασία πιο συντονισμένη και εποπτική. Με βάση λοιπόν αυτή την πρόσφατη επίσκεψή μου μπορώ να πω ότι φαίνεται να κατανοούν οι εταίροι μας ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουμε τον υφιστάμενο διάλογο. Και επίσης το εξήγησα, ε, ότι αυτό δεν είναι μια απόπειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπονομεύσει την ομοθεσία dot Frank. Τέταρτος τομέας, ε, η Ένωση Χρήματα Αγορών, το συζητήσαμε τον περασμένο μήνα, δεν θα το επαναλάβω, δεν θέλω να προσθέσω πολλά σε αυτή τη συζήτηση, απλώς να πω ότι ε, ανακεφαλαιώνοντας, η Ένωση Κεφαλαιογορών τι σημαίνει να συνδέονται οι αποταμιεύσεις με την ανάπτυξη. Θέλουμε λοιπόν να σπάσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν άμεσα στα χρήματα των επενδυτών και τις ευκαιρίες επενδύσεων για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που εμποδίζουν εκείνους που χρειάζονται χρηματοδότηση από το να φτάσουν στους επενδυτές. Και το σύστημα ε, για να διοχετευτούν αυτά τα κονδύλια, δηλαδή η αλυσίδα επενδυτική, θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Εάν τα καταφέρουμε και το στήσουμε σωστά, ε, θα μπορέσουμε να εθαρρύνουμε μακροπρόθεσμη επένδυση, επένδυση σε υποδομές και εναλλακτική χρηματοδότηση και επενδύσεις στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περιμένω να ακούσω με ανυπομονησία τις απόψεις σας, αλλά και των κρατών μελών, εθνικών κοινοβουλίων, ΜΚΟ, μικρομεσαίων και ε, του κλάδου. Έχουμε πάει με το επιτελείο μου μέχρι τώρα σε νέα κράτη-μέλη και προτιθέμεθα να πάμε και σε άλλα, στο υπόλοιπο της διαβούλευσης, με χαρά. Ε, ε, θα, θα μου να με καλέσετε κι εσείς αν κάνετε στα κράτη-μέλη σας τέτοιες εκδηλώσεις για ε, την ε, και την αναθεώρηση της οδηγίας για το χειρίδιο προσπέκτους. Ε, ε, ο στόχος μου θα είναι να γίνει πρόοδος όσο γίνεται πιο σύντομα και να προωθήσω νομοθετικές προτάσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Πέμπτη προτεραιότητα είναι να διερευνήσουμε πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερο ωφέλη άμεσα στους πολίτες, ωφέλη της εσωτερικής αγοράς. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλά για να διαδοθούν ε, ευεργετήματα από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να ταυτιστούμε με τους καταναλωτές και να δούμε ποια είναι τα εμπόδια ε, για για καλύτερο ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, ε, σε διασυνοριακά επενδυτικά ταμεία που έχουν διαφορετική επιβάρυνση για τη ε, λειτουργία τους, ε, τα τέλη δηλαδή. Ξέρουμε ότι ορισμένα ε, χρηματοπιστωτικά προϊόντα διαφέρουν στην τιμολόγησή τους από χώρα σε χώρα. Τους επόμενους μήνες λοιπόν θα ξεκινήσω μια διαβολεύση για να δω ποια είναι τα εμπόδια και πώς θα βοηθήσουμε τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα προϊόντα, καλύτερες υπηρεσίες και πιο φθηνές τιμές διαβούλευση για την Ένωση Αγορών θέλει να τονίσει και τις ε, λιανικές επενδύσεις και την ε, εμπιστοσύνη των ε, επενδυτών τη θεωρεί κλειδί και κεντρική ιδέα. Και επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί η γνώση των πολιτών για αυτά τα θέματα. Τα τελευταία χρόνια εγκρίθηκε πολύ μεγάλη νομοθεσία για τα χρηματοπιστωτικά ε, και σε δύσκολες συνθήκες και με χρονική πίεση και κανείς δεν το γνωρίζει καλύτερα από εσά, επιτροπή σας. Αυτή η ρύθμιση όμως και η νομοθεσία μας έδωσε ένα σύστημα πιο σταθερό και πιο ανθεκτικό. Εκτός από αυτό, νομίζω θα ήταν μια καλή ιδέα να δούμε αν υπάρχουν τίποτα ανεπιθύμητες συνέπειες και ποιο θα είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα αυτών των κανόνων. Καλωσορίζω την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής σας για αυτό το θέμα και προσβλέπω σε περαιτέρω συζητήσεις μαζί σας εν ευθέτω χρόνο. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όπως αναμένεται, θα κοιτάξουμε τους διάφορους νόμους ε, που περνούν με διάφορες ρήτρες αναθεώρησες που έχουν μπει σχεδόν σε όλα τα νομοθετήματα και θα πρέπει να το δούμε από πλευράς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αλλά και γενικότερα από πλευράς απασχόλησης και ανάπτυξης. Γενικότερα όμως θέλω να καταλάβω πώς επηρεάζουν οι κανόνες και οι πράξεις μας τα διάφορα νομοθετήματα και πώς βρουν ε, ε, το ένα μαζί με το άλλο. Δεν αφισβητώ καθόλου αυτέ τι μεταρρυθμίσει που χρειάστηκαν κόπο, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ σημαντική για εσά και η αναλογικότητα και στα δικά σα μάτια. Και ξέρω πόσο σημαντικέ είναι οι τη εργασία και η ανάπτυξη για όλους τους ε, ψηφοφόρου σα. Χαίρομαι ε, που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και προσβλέπω στις ερωτήσεις σας όχι μόνο σήμερα αλλά και τους επόμενους μήνες καθώς επιδιώκουμε να διατηρήσουμε τη χρηματοοικονομική σταθερότητα με τρόπο που να ευνοεί και ε, τις εργασίες και την ανάπτυξη αλλά και να εθαρρύνει την μακροπρόθεσμη επένδυση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε Χίλ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω τη συζήτηση. Πρώτος ομιλητής από το ΕΛΚΑ Κούτμαρ Χόκμαρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να σε ευχαριστήσω και εσάς κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση σας αυτή Προφανώς είστε πρόσδεκτος στην Επιτροπή μας και χαιρόμαστε πάντα να ακούμε τις ιδέες σας και τις συμβουλές σας για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον και είναι θετικό να ακούμε και κάποια σχόλια για το τι ήδη έχουμε κάνει και τι ήδη έχουμε πετύχει. Μία ερώτηση που ενδεχομένω να ακουστεί κάπως ηρωνική, πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που περιπλέκονται κάποια παλαιότερα project, σχέδια κτλ. Ξεκινάμε καινούρια. Πολλές φορές στα ίδια τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούμε μια νέα ένωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές διαφορετικές ενώσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες αυτές οι νέες ενώσεις ουσιαστικά σε τι αντιστοιχούν, στο ότι δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε εξ αρχής μια καλή Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να διορθώσουμε δηλαδή τα κακό κείμενα, τα προβληματικά σημεία που τομίσαμε στο παρελθόν, αποφασίζουμε να δημιουργήσουμε νέα σχέδια, νέα προγράμματα και το και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι χρειαζόμαστε απεγνωσμένα όλο και περισσότερες επενδύσεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τονίσετε κι εσείς ότι όντω χρειαζόμαστε νέε επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί νομίζω πραγματικά ότι αυτό είναι, αν θέλετε, η πρωταρχική προτεραιότητα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλέ συζητήσει γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το επενδυτικό σχέδιο, αλλά ξέρετε ότι πολλέ περισσότερε επενδύσει και πέρα από το επενδυτικό σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι γενικότερα πρέπει να ασχοληθούμε με όλο το χρηματοοικονομικό σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ λειτουργεί. Θα μπορούσατε λοιπόν να μα πείτε πρώτον πώ μπορούμε μέσω τη Ένωση Κεφαλαγορών να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία δεν καταφέραμε να πετύχουμε μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ θα γίνει αυτό στην πράξη. Και δεύτερον, πώς θα καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τα παλαιότερα προγράμματά μας, τα παλαιότερα θεσμικά προγράμματα, τους παλαιότερους θεσμούς, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οικονομία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρατούν κυρίως οι τράπεζες, οι οποίες επηρεάζουν τελικά ακόμα και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερων επιχειρήσεων πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι ίδιες οι τράπεζες θα αρχίσουν να καταβάλουν αυτές περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον καλύτερο, τον υψηλότερο δυνατό αριθμό επενδύσεων, να καταφέρουμε και να πετύχουμε βέβαια νέα επιτεύγματα, αλλά να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε και τα παλαιότερα προγράμματά μας. Ευχαριστώ. Well, I, um, I agree with you. Συμφωνώ μαζί σας. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι με την Ένωση Αγορών προσπαθούμε να επιτύχουμε στόχους που είχαμε θέσει και παλιότερα. Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, για παράδειγμα. Αυτό ήδη υπάρχει από τη συνθήκη της Ρώμης. Αλλά προκειμένου να καταφέρουμε να δώσουμε μια νέα στην οικονομία και μια πολιτική ακόμα όθηση στην οικονομία και να βασίζεται αυτή την πραγματική οικονομική ζήτηση και προκειμένου να καταφέρουμε να δούμε αν θέλετε και τα παλαιότερα προγράμματά μας, πρέπει να δούμε αν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Ή καταλαβαίνετε ότι μερικές φορές προκύπτουν εκτάκτως κάποια προβλήματα, τα οποία καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα και ενδεχομένω μέσω νέων προγραμμάτων. Συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ε, θα πρέπει να διατηρούμε μια απολογητική στάση κάθε φορά που εγκαταλείπουμε κάτι το οποίο κάναμε στο παρελθόν ή όταν επιστρέφουμε πολλές φορές σε κάτι το οποίο υπήρχε στο παρελθόν προκειμένου να το διορθώσουμε. Όσον αφορά τη διασύνδεση στην οποία αναφερθήκατε ανάμεσα στι κεφαλαγορέ, την Ένωση Κεφαλαγορών και τι τράπεζε, είναι πάρα πολύ σωστή. Προφανώ υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Η Ένωση Κεφαλαγορών δεν αποτελεί απειλή για τι τράπεζε, ούτε θα πρέπει να θεωρηθεί ω απειλή από τι τράπεζε. Νομίζω ότι έρχεται να συμπληρώσει το τραπεζικό τομέα και η ανταπόκριση που είχα μέχρι στιγμή από του εκπροσώπου του τραπεζικού τομέα σε διάφορα κράτη-μέλη ήταν γενικά θετική. Αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε όσον αφορά το τραπεζικό τομέα είναι σε ορισμένες ε, περιοχές, σε ορισμένες ε, πλευρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταφέρουμε να έχουμε την κατάλληλη ρύθμιση όσον αφορά τα τραπεζικά ζητήματα. Αυτό προσπαθήσαμε να πετύχουμε μέσω της οδηγίας και του κανονισμού για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Μπορούμε εκ νέου να εξετάσουμε όλες αυτές τις απαιτήσει και να διασφαλίσουμε τελικά ότι οι τράπεζες στα πλαίσια των κεφαλαγορών θα καταφέρουν να λειτουργούν θετικά. Για παράδειγμα, όσον αφορά την τυπλοποίηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια απλή διαφανή τυπλοποίηση επιτέλους. Αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό και για τις αγορές και για τις τράπεζες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αγορές και τράπεζες αλληλοσυμπληρώνονται και νομίζω ότι έχουμε πλέον την υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για να σημειώσουμε πρόοδο. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστές η κυρία Νίνα Τζίλ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ επίση για το είσαι για το MMF και πραγματικά θέλουμε μια έντονη δέσμευση από εσά προκειμένου να ασκήσετε πίεση στην Λετωνική Προεδρία για να προχωρήσει περισσότερο με το φάκελο αυτό. Ήταν λίγο διστακτική νομίζω στην αρχή και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια γενική τοποθέτηση του Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε και εμεί το συντομότερο δυνατό όταν ψηφίσουμε την έκθεση αυτή τον επόμενο μήνα στο Λομέλη θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε τριμερή διάλογο. Συμφωνώ επίση μαζί σα ότι πολλέ φορέ η εφαρμογή των διαφόρων οικονομικών νομοθετημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει ένα κάποιο κατακαιρματισμό. Ξέρω ότι ε, η κατάσταση διαφέρει από το ένα κράτο μέλο στο άλλο και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να διορθωθούν προτού προχωρήσουμε σε μια πραγματική ένωση κεφαλαγορών. Όσον αφορά την Ένωση Κεφαλαγορών, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα. Το να περιμένουμε μέχρι το 2019 για να αρχίσει να λειτουργεί η Ένωση αυτή, τη στιγμή που η οικονομική ε, ανάπτυξη στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ μικρή, η ενεργία είναι τεράστια. Καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε τώρα και επιγόντω την Ένωση Κεφαλαγορών. Τώρα χρειαζόμαστε τι επενδύσει ιδίω αν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε και του καταναλωτέ και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και πρέπει να ασχοληθούμε και με το ζήτημα τη διαφάνεια. Ξέρετε ότι ε, προσπαθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη δανειοδότηση. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να θεσπίσει μητρώα δανειοδότησης που ενισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ζήτημα επίσης της τιτλοποίησης. Όπως είπατε και εσείς, χρειαζόμαστε μια τυποποιημένη, απλή και διαφανή τιτλοποίηση. Ένα πολύ σημαντικό νέο εργαλείο στα πλαίσια της Ένωσης Κεφαλαγορών. Επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι η ομάδε πίεση στα πλαίσια των κεφαλαγορών θέλουν να έχουν όλο και λιγότερε απαιτήσει όσον αφορά τις, τα κεφάλαια, τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αυστηροί με τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει και να υπάρχει και απαραίτητη διαφάνεια. Διαφάνεια ιδίω κάθε φορά που υπάρχουν συναλλαγέ οι οποίε μεταφέρουν κίνδυνο από τον έναν τομέα στον άλλον. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και στο ζήτημα της μεταβίβασης, της διαβίβαση των δανείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς όλα αυτά θα μπορούσε να υιοθετήσει μια πρόταση που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα workshop, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα non-profit depository, ένα αποθεματικό ταμείο, το οποίο θα μπορούσε να ασχολείται με τα ζητήματα αυτά και με τα ζητήματα της έκθεσης σε υψηλό κίνδυνο από τραπεζικούς αλλά και μη τραπεζικούς φορείς στις οικονομικές αγορές. Κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω θα καταφέρουμε να αποφύγουμε και τη δημιουργία φούσκας στις κρεματαγορές. Κοιτάξτε, θα ήθελα να τονίσω, όπως είπα και στην Προεδρία, ότι όταν ήμουν στη Ρήγα προηγουμένως, τόνισα ότι μπορεί να βρούμε τρόπο πρόοδου και θα το ξανατονίσω και τώρα. Συμφωνώ με αυτό που είπατε γενικά για τη σημασία της εφαρμογής. Βασικά θεωρώ ότι θετήσει, αν νομοθετήσετε πρέπει να διασφαλίσετε και τη σωστή εφαρμογή και δίκαια και ισότιμη. και για την νομισματική ένωση, την ένωση των κεφαλαίων. Συμφωνώ, συμφωνώ. Είναι επίγον θέμα. Γενικά φροντίζω να δω τι μπορώ να κάνω με τις επενδύσεις, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Γενικά θέλω να βρω πάση θυσία τρόπο να το πετύχω γιατί αντιμετωπίζουμε συλλογικά αυτή την πρόκληση, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Και αυτή είναι η δουλειά μου, να σηκώνομαι κάθε πρωί και να βρίσκω τόπους, ιδέες. Συμφωνώ ότι είναι κατεπήγον και υπάρχουν βέβαια δύσκολες πτυχές, θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να καταλήξουμε κάπου, αλλά πρέπει να αρχίσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ενώ ταυτόχρονα θα κάνουμε την αναθεώρηση της ε, εξασφάλισης και θέλω και εγώ να γίνει πρόοδος σε όλους τους τομείς, όποτε γίνει δυνατόν. Και ελπίζω να έχω και την συνδρομή της Επιτροπής σας διότι έχουμε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να κάνουμε μια πρόοδο και πρέπει να την αδράξουμε. Τέλος για τη διαφάνεια συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα για τη σημασία που έχει η διαφάνεια και όλα όσα είπατε. Η διαφάνεια είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο και πρέπει να το προωθήσουμε. Ευχαριστούμε για να σεβαστούμε το χρόνο μας πρέπει ο καθένας να σέβεται και τα πέντε λεπτά. Αλλά αν πάρετε βέβαια συνολικά, γιατί αν πάρετε τρία λεπτά για την ερώτηση θα μείνουν μόνο δύο για την απάντηση. Και η Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίσατε Λόρδε Χίλ. Πολλές φορές έχω ασχοληθεί με το θέμα της κεφάλαια αγοράς Και τους τελευταίους δύο μήνες τουλάχιστον το συζητούσαν με όλοι. Το πρόβλημα μου είναι ότι συνήθως στα, στις μισές συνεδριάσεις μιλάμε για τις διαφορές και μετά για πτυχές του ΜΕΦΙΤ, του CSR e και άλλες τμηματικές νομοθεσίες ώστε φροντίζουν να μην μπορέσει να εφαρμοστεί ποτέ η Ένωση των Κεφαλαιαγορών. Οι σημερινές μας συζητήσεις με την ΕΣΜΑ και την Κομισιόν μας έδειξαν ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί το εξής, ιδιαίτερα ως προς τη διαφάνεια. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της διαφανείας, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα για την αγορά των ομολόγων. Γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η πιο ρευστή αγορά ομολόγων και δεν πέτυχαν να πετύχουν η χνηλασιμότητα παρά αποστεριόρια. Το επίπεδο 1 του ΜΕΦΙΤ το αναγνωρίζει αυτό και είναι φανερό ότι πρέπει να φροντίσουμε ιδιαίτερα το θέμα των κρατικών ομολόγων. Κάναμε μάλιστα συγκεκριμένες αναφορές στο ΜΕΦΙΤ, το τονίσαμε και στην ΕΣΜΑ ότι πρέπει να δούνε κατά πόσον είναι ελληνικοί ή χονδροπολιτές. Επίσης βάλαμε και άλλα πολλά κριτήρια για τα διάφορα χαρακτηριστικά της αγοράς ομολόγων. Το σημερινό μου λοιπόν ερώτημα είναι συμμερίζεστε την ανησυχία μου για την πιθανή διατάραξη που μπορεί να επιφέρει στις αγορές ομολόγων η πληροφόρηση μόνον εξ post και πώς θα μπορέσουμε τελικά να σταθμίσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να μην καταλήξουμε σε αυτήν την διατάρξη. Το ερώτημά σας ε, αφορά το κύριο ακριβώς θέμα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ και οι υπηρεσίε μου. Πώς να μπορέσουμε δηλαδή να σταθμίσουμε όντως σωστά, να εξισορροπήσουμε τη διαχείριση του κινδύνου με τρόπο που να μην υπερβολικά τουλάχιστον μειώνει την ανάπτυξη. Το πρόβλημα το γνωρίζω πολύ καλά όποτε σκέφτομαι την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών μου τίθεται. Η διαφάνεια λοιπόν που ζήτησε το ΜΥΦΙΤ είναι κάτι σημαντικό και το δεχόμαστε. Βέβαια πρέπει να ζυγιαστεί σωστά με τα εφαρμοστικά μέτρα γιατί δεν θέλουμε να βλάψουμε την ρευστότητα των κεφαλαίων Φυσικά εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να βλάψω τη λειτουργία της αγοράς ομολόγων και ξέρω ότι αυτό το θέμα σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα όπως και άλλους. Το ΕΣΜΑ όπως ξέρετε το συζητάει, το εξετάζει αυτή τη στιγμή. Είμαι βέβαιος ότι θα σκεφτούν και αυτοί αυτά που είπατε και εσείς και άλλοι και πιστεύω ότι και εγώ και οι υπηρεσίες μου θα βρούμε την κατάλληλη λύση αλλά πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα ώστε να έχουμε τελικά ένα σωστό σύγχασμα. Ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους ήταν Γέντζακ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Και εγώ με τη σειρά μου σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε για τα money market funds τα ταμεία χρηματαγορών και έχω την εξής ερώτηση. Πρόσφατα ακούσαμε ότι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες περιπλοκές ε, όσον αφορά το κρατήδιο της Καρινθίας που έχει μια εγγύηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπάρχει όμως μια ειδική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία οι κρατικές εγγύησεις θα μπορούσαν ε, να θεωρηθούν ε, μη ισχύουσες. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ε, νομική δράση που θα μπορούσε να ληφθεί. Αν όντως δεν ισχύσει η εγγύηση αυτή, τότε τελικά αυτό βάλει κατά τις οδηγίες για την ανάκαμψη των τραπεζών Δηλαδή θα πρέπει οι πιστωτές τελικά να αναλάβουν το βάρος ή θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι. Ποια είναι η στάση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στην πράξη πώς θα επηρεαστεί η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίαση των τραπεζών. Θα, θα τροποποιούσατε εσείς το BRRD, την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίαση σε, σε ένα τέτοιο σενάριο. Σας ευχαριστώ που θέσετε το ερώτημα αυτό και εν γένει, όσον αφορά την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση. Νομίζω ότι όντως θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος προκειμένου να μεταφερθεί σωστά στα κράτη-μέλη. Μετά τις μεταρρυθμίσεις που γίνανε κατά την προηγούμενη μας εντολή, το σύστημα είναι συλλογικά πολύ πιο ισχυρό από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία αναφερθήκατε, είναι μια περίπτωση πολύ πολύπλοκη και όντω εμπλέκονται παλαιότεροι και νέοι κανόνες και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί ότι η μεταβατική περίοδος από το ένα σύστημα στο άλλο ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποιες περιπλοκές. Για να απαντήσω πάντως στην ερώτησή σας, για το τι κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να σας πω ότι είμαστε σε στενή επαφή με τις Αυστριακές Αρχές. Δεν έχουμε στα χέρια μας όλες όμως τις πληροφορίες προκειμένου να καταφέρουμε να δώσουμε πλήρεις απαντήσεις. Πάντως, στα πλαίσια μιας προκατακτικής έρευνας που έχει γίνει, φαίνεται ότι η εφαρμογή του BRRD όπως έγινε από την Αυστρία την 1η Μαρτίου ήταν, απαραίτητη, ήταν δικαιολογημένη. Εφαρμόζονται λοιπόν οι κανόνες. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε αυτή τη στιγμή στο συμπέρασμα ότι πρέπει να τροποποιήσουμε την οδηγία ευθύ αμέσω. Αντίθετα θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην περίπτωση αυτή. Σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρη πάντως η περίπτωση αυτή, είναι αρκετά πολύπλοκη. και ξέρετε ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε περισσότερο εφόσον έχετε μάλιστα και ερωτήσεις τις επιπτώσεις του Μπέιλιν όσον αφορά τις γερμανικές τράπεζες. Μικέλ Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μία γενική ερώτηση και μία πιο συγκεκριμένη. Οι περισσότεροι θέλουμε προφανώ να πετύχουμε μια σταθερότητα όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα μπορούσατε εσείς να κάνετε έναν απολογισμό όπου να γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στις τραπεζικές δραστηριότητες όπου υπάρχει πολύ μεγάλη κερδοσκοπία να δούμε επίσης ποια διάκριση μπορεί να γίνει ανάμεσα σε εμπορικές και τις λιανικές τράπεζες Θεωρήθηκε διαχωρισμό αυτό πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια τη κρίση, αλλά δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι έχουν γίνει σπουδαία πράγματα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι πολύ μεγάλοι χρηματοοικονομικοί κολοσσοί, οι οποίοι δεν μπορούν να καταρρεύσουν και δεν πρέπει να καταρρεύσουν. Έχουμε το Ταμείο Εξυγίανση, το οποίο αντιστοιχεί μόνο στο 4% του ποσού που χρησιμοποιήθηκε για να ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζε. Αρκεί λοιπόν το ταμείο αυτό, μας καθησυχάζει μήπως πάλι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα καταβάλουν σημαντικό τίμημα. Επίσης, εποπτεία απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή τη στιγμή πέρα από την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής θα είναι σε θέση να αποκριθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις νέες αυτές αρμοδιότητες. Επίσης, ξέρετε ότι 4 δισεκατομμύρια δολάρια χρειάστηκε να καταβληθούν από έναν συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό οργανισμό στι ΗΠΑ, επειδή ουσιαστικά είχε παραπλανήσει του πελάτε του. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε όλο και περισσότερο στο ρόλο που έχουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, στην ευθύνη που φέρουν, ιδίω όταν πρόκειται για οίκου αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Well, um, in, in reverse order, on credit ratings. Λοιπόν, όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα και την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, στα πρώτα ήμιση του 2015 θα έχουμε μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τους οίκους αξιολόγησης. Θα μας δοθεί τότε η δυνατότητα λοιπόν να εξετάσουμε περισσότερο τα θέματα που φίξατε. Όσον αφορά τώρα το πρώτο, την πρώτη σας παρατήρηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τραπεζικός τομέας και την κεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα, η δική μου άποψη είναι ότι, και το είπα αυτό και πριν από λίγο, εν γέννη οι τράπεζε βρίσκονται σε πολύ πιο θεκτική και καλύτερη στάση από ό,τι βρισκόντουσαν στο παρελθόν. Νομίζω ότι έχει γίνει μια σφαιρική αξιολόγηση, η οποία καταδεικνύει ότι οι τράπεζε είναι πλέον πολύ πιο αθεκτικές και στεναρέ και σταθερέ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν με αυτό. Και το Ταμείο Εξυγίανση έχει αρχίσει σιγά σιγά να δημιουργείται, να στείνεται. Επομένω, θα προέρχεται και από αυτό ένα μεγαλύτερο βαθμό ανθεκτικότητα για τι τράπεζε. Όσον αφορά το ζήτημα τη ανεξαρτησία, το οποίο αναφερθήκατε. Προφανώ η ανεξαρτησία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ο νέο υποπτικό μηχανισμό όντω προσδίδει στον μηχανισμό αυτό μία ανεξαρτησία όσον αφορά τη λειτουργία του. και όπως είπα και πριν από λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντική και η ποιότητα του προσωπικού που χρησιμοποιούμε στα πλαίσια του Συμβουλίου Νέας Εξυγένσης, ένα συμβούλιο το οποίο λειτουργεί ήδη καλά, έχει αρχίσει να εργάζεται, γνωρίζουν οι άνθρωποι στο Συμβούλιο αυτό ότι τους περιμένει μια τεράστια πρόκληση, θα αρχίσουν να λειτουργούν πλήρως από τον Ιανουάριο, αλλά έχω έρθει σε επαφή μαζί τους και συνειδητοποιούν αυτή τη στιγμή πόσο σημαντική είναι η αρμοδιότητά τους και είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτές τις νέες τους αρμοδιότητες. Ευχαριστούμε Μόρελ Σκότ από τους Πρασίνους. Βλέπουμε να ανησυχείτε ε, για τις μικρομεσαίες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Αλλά πάει καιρό τώρα ε, που δεν ε, επενδύουν στις μικρομεσαίες. Στην παλιά οικονομία ε, το παλιό πεθαίνει, αλλά το καινούριο δεν μπορεί να γεννηθεί. Οι νέοι τομεί χρηματοπιστωτική στο μέλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν για να έχουμε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων να προωθηθούν αυτέ τι επενδύσει. Οι τράπεζε δεν δίνουν τι επενδύσει που χρειάζονται οι μικρομεσαίε. Εμεί οι πράσινοι πιστεύουμε ότι έχει να βαγίσει ο κλασικό παραδοσιακό τραπεζικό τομέα γιατί δεν αποδίδουν και η τιτλοποίηση και κάποιες άλλες ε, κερδοσκοπικές δραστηριότητες των τραπεζών αποδίδουν περισσότερο. Ε, θα πρέπει λοιπόν περισσότερο να ρυθμιστεί η κλασική τραπεζική λειτουργία και να σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνουν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τρόπο προβλέψιμο και με ε, λογικά επιτόκια. Και αυτό γίνεται καλύτερα έτσι από τις ένας βασικός ρόλος που θέλουμε για τις τράπεζες και είναι κοινωνικός είναι η εκτίμηση κινδύνου, η εκτίμηση των, της πίστοσης σε στενή συνεργασία με τον πελάτη. Αυτό μόνο τράπεζα μπορεί να το κάνει. Και θέλω λοιπόν να σας παρουσιάσω μερικές ιδέες που έχουμε εμείς οι πράσινοι. Πρώτον, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις τράπεζες Λιανικής τη σχέση με τον πελάτη για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να υποστηρίζουν τις πιο παραγωγικές και πιο υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, ε, ε, διάφορα ε, μοντέλα τοπικά στις διάφορες τοπικές κοινωνίες να μπορούν να υποστηρίζουν και να επενδύουν στις δικές τους εταιρείες και αυτό σημαίνει και μεγαλύτερη λογοδοσία και πιο κοντά και πιο μικρές αποστάσεις για να μπορούν να έχουν διαφοροποίησει το πηγών τους, χρηματοδότηση εταιρείε. Και για να ενημερώνονται καλύτεροι επενδυτέ, μπορεί να υπάρχει και μια υπηρεσία αξιολόγηση του αξιόχρεου τη ίδια τη εταιρεία. Το είπατε και εσεί στην παρουσίασή σα. Θα πρέπει να δίνονται κίνητρα με πιο μακροπρόθεσμε επενδύσει, ποιοτικέ, είναι, έχουν μεγαλύτερη ένταση κεφαλαίου και λόγω του κινδύνου δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν ακριβώς σε τοπικό επίπεδο. Μια λογική απάντηση ήταν εξή. Αν υπάρχουν ειδικέ ιδέες που θέλετε να διερευνήσετε περισσότερο, για να μην σας δώσω τώρα απαντήσεις με επικεφαλίδες, καλό θα ήταν να το δούμε διμερώς. για να εξετάσουμε ενδεχομένω ε, πού μπορούν να ενταχθούν οι ιδέες αυτές. Η γενική μου άποψη θα ήταν η εξή. Προσπαθώ να βοηθήσω να πετύχουμε με την ένωση των κεφάλαιων αγορών είναι το εξή. Να έχουμε διαφοροποιημένο σύστημα. Είναι γεγονός ότι οι τοπικές τράπεζες που έχουν και τοπικά δίκτυα και σχέσεις ε, εργάζονται καλά και συνεργάζονται με τις εταιρείες οι οποίες παίρνουν τα χρήματα που τους χρειάζονται ως πιστώσεις για να λειτουργούν. Αλλά εξεπλάγει πάρα πολύ όταν μιλούσαμε με κάποια πιο νέα κράτη-μέλη που είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι στις χρηματαγορές τους και λιγότερο ανεπτυγμένη επιχειρηματική παράδοση και τους άρεσε η χρηματοδότηση εκεί από κεφάλαια. Το πρόβλημα είναι όταν βάζεις όλα σου τα αυγά στο ίδιο καλάθι, μπορεί να σπάσουν. Mm αν έχεις μια οικονομία που εξαρτάται πάρα πολύ ισχυρά από τη χρηματοδότηση των τραπεζών και υπάρχει κάποια στιγμή μια σύσπαση, ένα πρόβλημα στη λειτουργία των ε, τραπεζών, αυτό έχει τεράστια επίπτωση στην οικονομία. Και εν μέρει αυτό συνέβη στην ευρωπαϊκή οικονομία τα τελευταία χρόνια. Αυτό που επιδιώκω εγώ λοιπόν και με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι μια διασπορά ε, πηγών χρηματοδότησης τέτοια ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις και να έχουν πρόσβαση σε διάφορα στάδια ανάπτυξής τους. Στα κεφάλαια κινδύνου δεν είμαστε καλοί παντού στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις νεοφύης που ξεκινάνε και μετά πηγαίνουν στις ΗΠΑ για να χρηματοδοτηθούν και να αναπτυχθούν ας πούμε ε, νέες καινοτόμες ε, εταιρείες ε, high-tech και πηγαίνουν γιατί είναι πρόσφορο το έδαφος και το περιβάλλον. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ευελιξία και κίνητρα για πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις και στις υποδομές έχει σημασία και εγώ θέλω πολύ να το προωθήσω αυτό. Thank you. I Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ πολύ δύο λεπτά μόνο για τις ερωτήσεις σας. Ο κύριος Τζάνι για το EFDD, ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις για τον Επίτροπο. Πρώτη, μια γενική ερώτηση όσον αφορά την Ένωση Κεφαλαγορών. Εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσατε λοιπόν την πράσινη βίβλο σας, παρουσιάσατε τις παρατηρήσεις σας, παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με το ότι η Ένωση Κεφαλαγορών τελικά θα βοηθήσει, λέτε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του παραγωγικού ευρωπαϊκού συστήματος. Η μεγάλη όμως αμφιβολία που τίθεται και που έχω εγώ και που δεν νομίζω τελικά ότι θα επιτευχθεί μέσω της Ένωσης Κεφαλαγορών είναι πώς θα καταφέρουμε να συμφιλιώσουμε τα συμφέροντα των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών με τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να συμφιλειωθούν αυτά τα δύο, αυτά τα δύο συμφέροντα. Και πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένω να οδηγηθούμε σε μία εκ νέου επαναχρηματοδότηση ή την έλλειψη μάλλον χρηματοδότηση, με συγχωρείτε, της ε, ε, πραγματικής οικονομίας. Ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τώρα την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίαση των τραπεζών και όσον αφορά γενικότερα την Τραπεζική Ένωση. Θα πρέπει προφανώς να αρχίσει να εφαρμόζεται η οδηγία αυτή αλλά ενδεχομένως οι επιπτώσεις της οδηγίας αυτής να μην αρκούν για να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα που έχουμε στο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ευρώπη. Η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση ουσιαστικά θα λειτουργήσει για τις επιπτώσεις που έχουμε στα πλαίσια μιας συστημικής κρίσης, αλλά δεν θα θεραπεύσει τη ρίζα του προβλήματος. Ξέρετε ότι είχαμε κάποιες μικρές τράπεζες στην Ιταλία, την ΕΤΑ, την Ελ οι οποίες ε, ουσιαστικά εξαρτώνται πάρα πολύ από τον τρόπο που λειτουργούν άλλες τράπεζες και πολλές φορές η ε, δική τους η πτώχευση βοήθησε τράπεζες ξένες όπως οι γερμανικές. Θα μπορούσαμε στα πλαίσια της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίαση των τραπεζών να έχουμε έναν πραγματικό διαχωρισμό στο οικονομικό σύστημα της Ευρώπης προκειμένου τραπεζικός τομέας πραγματικά να υποφελεί την πραγματική οικονομία. Κοιτάξτε, η δική σας Επιτροπή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ασχολείται με το ζήτημα της διάρθρωσης τραπεζών. Πολύ περισσότερο από ό,τι οποιοδήποτε άλλος και στην Ευρώπη θα έλεγα. Συνεπώς, έχετε μπροστά σας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή θα καταφέρει να μας προστατεύσει ακόμα περισσότερο από, τις, από τους μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι θεωρούνται too big to fail, πολύ σημαντικοί για να καταρρεύσουν ή θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε περισσότερο πώς λειτουργούν κάποιοι πολύπλοκοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Συμφωνώ πάντως μαζί σας ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις όσον αφορά την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση, την οδηγία BRRD. Βρισκόμαστε ακόμα στην ε, απαρχή της οδηγίας αυτής. Θα πρέπει καταρχάς να μεταφερθεί επαρκώς σε όλα τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια προφανώς να τεθεί σε ισχύ πανευρωπαϊκά. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, όπως γίνεται κάθε φορά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φορά που μεταφέρουμε οδηγίες προσπαθούμε να συνοδεύονται οι οδηγίες αυτές από τα απαραίτητα εκτελεστικά μέτρα προκειμένου να εφαρμόζονται πλήρως. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η βασική μου προσέγγιση είναι να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά διαφορετικά ζητήματα, τα οποία ενδεχομένω να περιπλέκουν αυτή τη στιγμή την πρόσβαση σε δανειοδότηση από μικρομεσαίες επιχειρήσεις δανειοδότηση την οποία χρειάζονται προκειμένου να εξελιχθούν, να αναπτυχθούν. Δεν μπορώ να δώσω μία και μοναδική λοιπόν απάντηση στο πρόβλημα. Μία πτυχή του προβλήματος είναι πώς θα καταφέρουμε να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία, αν θέλετε, πραγματική βιομηχανία, έναν κλάδο επιχειρηματικού κεφαλαίου, κεφαλαίου κινδύνου, πώς θα καταφέρουμε να έχουμε ε, περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς εν τέλει θα καταφέρουμε να πείσουμε και άλλους επενδυτές, πέρα από τους σημαντικούς και τους βασικούς, να επενδύσουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι δεν πρόκειται να επενδύσει κανείς αν δεν έχει μια κάποια προβλεψιμότητα, μια κάποια ενημέρωση όσον αφορά τον κίνδυνο. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν που συζητήσαμε είναι πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες πληροφορίες όσον αφορά τις πιστώσεις, προκειμένου οι επενδυτές να γνωρίζουν πραγματικά σε τι επενδύουν. Η απάντηση λοιπόν δεν είναι εύκολη. Δεν μπορούμε απλώς να πούμε ότι οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να ασχοληθούν με, τον, με τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ανταυτού θα πρέπει να έχουμε μια μεγάλη γκάμα, ένα μεγάλο φάσμα δανειοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό θα βοηθήσει εν γέννη και την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λόρδε Χίλ, πριν από ένα μήνα περίπου μας παρουσιάσατε την πράσινη βίβλο σας εδώ στην Επιτροπή για την Ένωση Κεφαλαίου Χωρών. Σας είπαμε. Μάλλον είπατε ότι θέλετε να ρίξετε τα εμπόδια βαθμιαία και σταδιακά για να βοηθήσετε για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το είπατε και σήμερα. Θα πρέπει να έρθουν ε, κοντά οι καταθέσεις, οι αποταμιεύσεις με τις ε, επενδύσεις ε, σε εταιρείε για δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θέλω να μπω σε δύο πράγματα. Καλύτερη πρόσβαση σε ανεξάρτητες ε, και διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Είπατε ότι το venture ε, capital, το κεφάλαιο κινδύνου του επιχειρηματικού είναι πολύ σημαντικό. Είδατε την έκθεση της Sands και Young που λέει το 2014 διεθνώς ε, ανθούσε πάνω από 86 δισεκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια έχουν επενδυθεί στο κεφάλαιο αυτό 60% στις Ηνωμένε Πολιτείε τα μισά από αυτά στο Silicon Valley, 12% στην Κίνα και 18% συγγνώμη, και μόλις 12% στην Ευρώπη. Τι θα κάνετε λοιπόν έτσι ώστε να προσελκύσετε και να ενισχύσετε αυτή την αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ευρώπη. Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να σας δώσω μια σωστή απάντηση και λογική. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε ε, το κεφάλαιο κινδύνου και τις αντίστοιχες αγορές να αναπτυχθούν στην Ευρώπη. Διότι και μόνο το γεγονός ότι βλέπουμε ευρωπαϊκές εταιρείες συνεχώς να μετεγκαθίσταται για να αντλήσουν ε, μάλλον χρηματοδότηση από το εξωτερικό, αυτό δεν είναι καλός ιονός για το μέλλον της οικονομίας μας και την ανάπτυξή της. Βεβαίως Υπάρχει ανάγκη να τονωθεί. Ο στόχος τώρα ποιος είναι των διαβουλεύσεων της, λευκής, της ε, πράσινης συγγνώμη, βίβλου. Είναι να δούμε όλους τους ενεχομένους, εκείνους που εργάζονται σε αυτά τα κεφάλαια κινδύνου ή άλλους, κράτη-μέλη, ξέρω εγώ, κοινωνία των πολιτών, να μας δώσουν όλοι τις ιδέες τους για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, αν υπάρχουν ειδικά εμπόδια που μπορούμε να ξεπεράσουμε, ποια βήματα ενδεχομένω να χρειάζεται να κάνουμε. Στην περασμένη θητεία νομίζω, η Ιουβέκα και η Ιούσεφ ήταν ε, κάποια νέα στοιχεία που εισήχθησαν. Ξέρω ότι έγινε κάποια πρόοδος και άλλα ταμεία ε, δημιουργήθηκαν. Θα πρέπει να το δούμε αυτούς τους κανονισμούς, δηλαδή να τους μελετήσουμε εάν και κατά πόσο λειτουργούν προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε εμείς και αν βοηθούν έτσι ώστε τα κεφάλαια κινδύνου και η κοινωνική χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση της κοινωνικής ε, επιχειρηματικότητα σαν συνάδων. Εγώ είμαι πρόθυμος να ακούσω προτάσεις, συστάσεις για το πώς μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Thank Ντανούτα Χούμπνερ. Η Ντανούτα Χούμπνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι πάρα πολύ που λαμβάνετε σοβαρά όλους αυτούς τους πυλώνες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, όχι μόνο τον πυλώνα της διαμεσαβο... διαμεσαλο... διαμεσολάβησης, με συγχωρείτε, αλλά και τον πρώτο πυλώνα που έχει να κάνει με τους προμηθευτές. Μπορείτε να μας πείτε σήμερα με κάποια σαφήνεια τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις αποταμιεύσεις προκειμένου να μην φεύγουν από τη δική μας την αγορά την ευρωπαϊκή σε τρίτες χώρες, αλλά πώς θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε και περισσότερες επενδύσεις και αποταμιεύσεις. Εν γέννη πιστεύετε ότι ε, μπορούμε να λάβουμε δράση μέσω ενός κανονισμού ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τις δυνάμεις που υπάρχουν στην αγορά, να εφαρμόσουμε κάποιες βέλτισες πρακτικές. Πιστεύετε ότι πρέπει να αναλάβουμε διαφορετική δράση, όχι αναγκαστικά μέσω κανονισμού. Και διατρέχουμε μήπως τον κίνδυνο να καταλήξουμε σε κάποια μέσα τα οποία τελικά θα διώξουν τις αποταμιεύσεις από τις δικές μας χρηματοπιστωτικές αγορές. Γιατί ελοχεύει και αυτός ο κίνδυνος. Πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Τώρα, όσον αφορά το FTT, δεν το αναφέρατε. Πάντως, στα πλαίσια της Ένωσης Κεφαλαγορών και το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό. Αναφερθήκατε στην ελεύθερη ροή κεφαλαίων. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας το τέλος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Τι θα γίνει ακριβώς με αυτό. Θα επέμβει για το ζήτημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί στα πλαίσια της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας κάπου έχει κολλήσει λίγο το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να λάβει δράση, θα κάνει κάτι γι' αυτό, να ξεχάσουμε εντελώ το τέλος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, το γενικότερο ερώτημά σας όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, τη χρησιμοποίηση κανονισμών ή όχι, η άποψή μου είναι ότι όπου απαιτείται νομοθεσία, τότε θα πρέπει να νομοθετούμε, όπως για παράδειγμα για τις τυπλοποίησεις ή για άλλα ζητήματα, τότε ναι, να νομοθετούμε, αλλά αν μπορούμε από την άλλη να πετυχαίνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς να νομοθετούμε αναγκαστικά, για παράδειγμα μέσω βέλτιστων πρακτικών, μέσω άλλων εργαλείων της αγοράς, τότε είναι υπέρ και αυτής της τακτικής. Και αυτό γιατί ξέρετε ότι απαιτείται πάρα πολύ χρόνο για να νομοθετήσει κανεί. Και συνάδει με αυτό που είπε η Νίνα Γκίλ, ότι πολλέ φορέ συναγκαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε έκτακτε καταστάσει. Αν λοιπόν μπορούμε να πετύχουμε σε ένα συγκεκριμένο τομέα πολλά πράγματα χωρί νομοθεσία και πολύ πιο γρήγορα, τότε εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορώ να υποστηρίξω με τέτοια προσέγγιση. Και εν γέννη, Όσον αφορά τα επόμενα στάδια στη δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαιογορών τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, πραγματικά νομίζω ότι θα έχουμε ένα μείγμα πολιτικής, μείγμα νομοθετικών και μη νομοθετικών προσεγγίσεων. Αυτά όσον αφορά το πρώτο ερώτημα. Όσον αφορά τώρα γενικότερα τις αποταμιεύσεις. Αυτό το οποίο ελπίζω είναι να έχουμε μία γκάμα μέτρων που θα καθιστούν πιο εύκολη και πιο ελκυστική τη δημιουργία μεγάλων κεφαλαγορών στην Ευρώπη, ότι θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερους επενδυτές. Ξέρετε ότι ε, πολλές φορές πέρα από τους μεγάλους επενδυτές έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν μόνο και μόνο για τα πιο όρημα χρόνια τους αν θέλετε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποταμιεύουν σε συγκεκριμένα ταμεία προκειμένου να καλύψουν τα χρόνια της ε, σύνταξής τους. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο αποτελεσματικά θα πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένες οι αγορές και θα πρέπει και επενδυτές να αισθάνονται ότι υπάρχει κατάλληλη ασφάλεια προκειμένου να επενδύσουν. Οι κεφαλαγορές λοιπόν προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά και να μην ενέχουν κινδύνους θα πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένες. Όσον αφορά το τέλος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο Επίτροπος Μοσκοβισή είναι αυτός που ασχολείται με το ζήτημα. Εγώ ανέκαθεν ναι, πίστευα ότι το ζήτημα αυτό είναι καλύτερα να το αντιμετωπίσουμε σφαιρικά διότι ζούμε σε έναν ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο ανταγωνιστικό κόσμο, θα πρέπει αυτό να το γνωρίζουμε ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα αυτό θα είναι να δώσει μια τεχνική υποστήριξη για τις χώρες εκείνες που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο με αυτή την πρωτοβουλία. Αυτό ήδη έχει γίνει και μάλιστα ο κύριος Μασκοβισή είπε πρόσφατα ότι θέλει να καταλήξει σε μια ρεαλιστική και φιλόδοξη συμφωνία τώρα όσον αφορά τη δική μου την άποψη. Νομίζω ότι οι επιπτώσεις που θα έχει ένα τέτοιο τέλος χρηματοπιστωτικών συναλλογών για την ένωση κεφαλαγορών, για την ανάπτυξη αλλά ακόμα και την απασχόληση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή σε μια ενδεχόμενη μελλοντική εφαρμογή ενός τέτοιου τέλους θα πρέπει και αυτές οι επιπτώσεις να τις λάβουμε υπόψη μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Και αυτό για λόγους κυρίως χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ποια είναι η αποψή σας για τα μέτρα αυτά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμφωνείτε με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεύτερον. Δεύτερον λέγω οι φραγμοί που τίθενται στις διαμεθοριακές επενδύσεις και εμποδίζουν τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως είπατε σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα, αν θέλουμε να στηρίξουμε καλύτερα την πραγματική οικονομία και μακροπρόθεσμα και τις υποδομές θα έπρεπε να προβλέψουμε επενδύσεις και από ιδιωτικά κεφάλαια και δημόσιες επενδύσεις, παραγωγικές όμως. Ενώ ξέρουμε ότι σε κάθε κράτος η διασύνδεση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων διαφέρει από κράτος σε κράτος και αυτό έχει διαφορετικά αποτελέσματα και επί της αγοράς. Έχετε μήπως τίποτε γενικότερο να μας πείτε γι' αυτό ώστε να υπάρχει ισονομία και ισοτιμία. Και τέλος, όπως ξέρετε, γιατί το είπαμε πολλές φορές, η Ένωση της Κεφαλαίου Αγοράς αφορά και τις τριτλοποίησεις και επομένως υπάρχει ο κίνδυνος να ξαναγνωρίσουμε τα ίδια προβλήματα που γνωρίσαμε πριν από μερικά χρόνια. Ενώ ξέρουμε ότι για να δουλεύει το σύστημα χρειάζεται εμπιστοσύνη των αγορών και όλων των αραγόντων. Πώς θα μπορούσαμε να πιστοποιήσουμε στου πολίτες ότι σήμερα έχουμε στοιχεία που να του προστατεύουν ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Σα ευχαριστώ. to take um, securitization first. Uh, um... Η τιτλοποίηση είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό στην ανάλυση μας. Γνωρίζουμε καλά τι συνέβη στο παρελθόν και δεν το θέλει κανείς αυτό. Ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ να ξαναγίνουν τα ίδια δηλαδή. Αυτό είναι σαφές ότι αυτές οι επικίνδυνες ρεψοκίνδυνες τιτλοποιήσεις δεν πρέπει να ξανάρθουν. Και νομίζω επομένως ότι, ότι λέγω πρέπει να προσέξουμε πώς, πώς λέγω, θα επιστρέψουμε με λογικό τρόπο σε τιτλοποιήσεις απλές και διαφανείς και τυποποιημένες. Με ενθαρρύνει το γεγονός ότι η Έκτη, η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας ή της ε, Βρετανίας, με συγχωρείτε, το προσέχουν επίσης και δεν πρόκειται εδώ για οργανώσεις που θέλουν να αναλάβουμε τέτοιους κινδύνους θα υπάρξει τρόπος. Αλλά αυτό με φρόνηση και με την υποστήριξη και συνεργασία ως το δυνατόν ευρύτερη και με εκπροσώπους της βιομηχανίας και φυσικά θα γίνουν διαβουλεύσεις μέχρι το τέλος Μαΐου και με τότε θα έρθουμε να κάνουμε προτάσεις νομοθετικές προτάσεις μάλιστα. Για την Ένωση των, της Κεφαλαίου Αγοράς, ένας από τους στόχους της είναι να αυξηθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το λέει η Πράσινη Βίβλος και αυτό. Υπάρχουν τρόποι και γι' αυτό για να είναι πιο ελκυστικές οι τιτλοποιήσεις ας πούμε ή και άλλοι τρόποι, άλλοι τρόποι ε, διατάξεις για τους ασφαλιστάς μέτρα δηλαδή που θα είναι πανενοσιακά και συνεπή για το πρώτο που είπατε για την ποσοτική χαλάρωση και γενικότερα την κατάσταση της οικονομίας Φυσικά, εγώ ασχολούμαι και με τη δημοσιονομική σταθερότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και πρέπει να γνωρίζουμε και τις μακροπροληπτικούς, μακροπροληπτικούς κινδύνους και τους μικροπροληπτικούς διούτους. Οι μάκρο λύνονται κυρίως μέσω του ESRP και πρέπει όπως ξέρετε φέτος να ξαναδούμε τις διευθετήσεις που θα κάνουμε για να δούμε αν χρειάζονται αλλαγές. Γενικά όμως νομίζω ότι φυσικά χρειαζόμαστε, πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, αλλά σίγουρα ο κύριος Τράγκη ο ίδιος το πράττει από την έκτο. Brian Hayes. Brian Hayes. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας τον uh, Επίτροπο Χίλ και συγχαρητήρια για το ότι έχετε ήδη πάει σε 9 κράτη-μέλη όπως μας είπατε. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εσάς και το γραφείο σας για τη διαθεσιμότητα σας αυτή, ότι πηγαίνετε πραγματικά και ακούτε τι έχουν να πούνε οι άνθρωποι, τι έχουν να πούνε οι καταναλωτές και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην uh, οικονομία. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με το TTIP. Νομίζω ότι είπατε ξεκάθαρα σήμερα ότι κάποια σχόλια που κάνετε στο Brooking Institute στις 23 Φεβρουαρίου, όπου αναφερθήκατε σε πραγματεύσεις αυτές, μιλώντας δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μας είπατε, ή είπατε τότε ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη συνεργασία από τη μία πλευρά που έχει να κάνει ουσιαστικά με τον ανεπίσημο διάλογο και με τις επαφές και συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη πλευρά ανάμεσα στους κοινού κανόνες που πρέπει να υπάρχουν. Μετά τον λόγο λοιπόν αυτό που εκφωνήσατε το Φεβρουάριο στις ΗΠΑ, τι ακριβώς προσπαθούμε εμείς να πετύχουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει στα πλαίσια του τύπη να υπάρχει και ένα κεφάλαιο ξεχωριστό που να έχει να κάνει με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τουλάχιστον θα πρέπει να πετύχουμε μια κοινή συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ξέρω ότι ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε προσεγγίζουν τα πράγματα διαφορετικά, θεωρώντα δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει μία και μοναδική δική του προσέγγιση όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα. Νομίζω πάντω ότι θα πρέπει να υπάρχει επαφή και στον τομέα αυτό, ακόμα και αν καταλήξουμε τελικά με δύο διαφορετικά καθεστώτα όσον αφορά τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ξέρετε ότι στο παρελθόν είχαμε σχετικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καταφέραμε τελικά να φέρουμε τις ΗΠΑ στη δική μας την πλευρά. Πώς πάνε διαπραγματεύσει για το ζήτημα λοιπόν αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς να σα ευχαριστήσω για τι γενικέ αυτέ παρατηρήσει σα και για το ότι ε, χαίρεστε κι εσείς από το ότι, ε, για το ότι επισκέπτομαι κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αποτελεί σημαντική αρμοδιότητα ενός ε, επιτρόπου αυτό, να έρχομαι σε επαφή δηλαδή με εκπροσώπους διαφόρων κρατών μελών και επιτόπου να ακούω ότι έχουν να πούνε οι πολίτες, οι οργανώσεις καταναλωτών, αλλά και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι επαγγελματίες δηλαδή αυτού του τομέα οφείλω εγώ ως Επίτροπος να γνωρίζω ότι έχουν να πούν οι άνθρωποι αυτοί για το, τον αντίκτυπο που οι αποφάσεις μας έχουν στην πραγματική οικονομία. Δεν μπορούμε λοιπόν να λειτουργούμε εμεί απομονωμένα από του ανθρώπου αυτού όσον αφορά τώρα το TTIP και τι Πολιτείες. Πώ έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι εσεί συνοψίσατε πολύ καλά τα πράγματα. Στόχος μας μέσω της επίτευξης μεγαλύτερης συνεργασίας στο χρηματοπιστωτικό τομέα για το TTIP έχει να κάνει με το ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ένας ιδιαίτερα ρυθμισμένος τομέας και μέσω της ρύθμισης αυτής ελέγχουμε τελικά και την πρόσβαση στις αγορές. Επομένως, το να έχουμε μια συμφωνία εμπορική, εμπορικών συναλλαγών, χωρίς να υπάρχει κεφάλαιο για το χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν είναι σωστό. Χάνουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Να ευχαριστήσω πάντως και τη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε μαζί, αν θέλετε, οι δύο ήπειροι αντιστοιχούν σε ένα, στο μεγαλύτερο τμήμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που έχουμε στον κόσμο. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων που πολλές φορές απορρέουν από παγκόσμια πρότυπα. Τις περισσότερες φορές τα πράγματα κινούν ομαλά, κινούνται ομαλά, αλλά άλλες φορές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των CCP, τα πράγματα δεν κινούνται ομαλά. Επομένως, ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα φόρα ρυθμιστικά που μας δίνουν τη δυνατότητα να συζητούμε τα ζητήματα αυτά. Δυστυχώς τα τεχνικά αυτά φόρα δεν είναι υψηλόβαθμα, είναι αρκετά ανεπίσημα και συνεπώς δεν γίνεται η συζήτηση στο κατάλληλο επίπεδο, αν θέλετε. Αυτό ακριβώς είπα λοιπόν στους ε, εταίρους μας, στις Ηνωμένε Πολιτείες, εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες. Σε καμία περίπτωση και τους καθησύχασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να επισέλθει στις δικές τους αρμοδιότητες. Το ζήτημα πάντως του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις ΗΠΑ, πάντως εμείς δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Θα προαφήσουμε δηλαδή τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Ο κ. Φερνάντες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Εγώ σας είχα τρεις ερωτήσεις και ελπίζω πολύ σύντομα να τις παρουσιάσω. Πρώτη, δεν έχει να κάνει με την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, αλλά με τα μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και εμείς που είμαστε εδώ βουλευτές, ή ε, ε, βοηθοί μας για να ανοίξουμε τραπεζικούς λογαρισμούς σε χώρες που δεν ζούμε, για να πληρώσουμε σε τράπεζες ξένες, τη μικρή καθημερινότητα που χρειάζεται βελτίωση για να μπορεί να λειτουργεί στο σύνολό της η νομισματική και η οικονομική ένωση. Και θα ήταν καλό να το σκεφτούμε αυτό. Μπαίνω λοιπόν τώρα στην πράσινη βίβλο αμέσω και έχω την εξή ερώτηση. Εγώ καταλαβαίνω ότι η Πράσινη Βίβλος θέλει να διευρύνει την γάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών που μπορούν να ε, χρησιμοποιούν ε, οι διάφοροι οργανισμοί πέραν των κλασικών τραπεζών. Οπότε η Πράσινη Βίβλος ποντάρει στην ανάγκη εναρμόνισης ε, των φορολογικών πλαισίων, των λογιστικών προτύπων ή ακόμα και τους νόμους για το πτωχευτικό δίκαιο. Στην Ισπανία έχουμε σοβαρά ελλείμματα στην νομοθεσία μας. Οπότε θα πρέπει να εναρμονίσουμε αυτό το σύστημα για να ε, μπορούν τα κεφάλαια να ρέουν αποτελεσματικά και να κατανέμονται. Εσείς πώς νομίζετε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχει και η δέσμευση του κυρίου Γιούνκερ να εναρμονίσει ε, ε, τη φορολογική βάση για το φόρο των επιχειρήσεων που συμβαδίζει με όλα αυτά που συζητάμε σήμερα. Και τελευταίο, πώς φαντάζεστε την ε, σύνδεση της Τραπεζικής Ένωσης με την Ένωση Κεφαλαιογορών, γιατί όλες οι χώρες που θα είναι στην Τραπεζική Ένωση δεν θα συμμετέχουν στην Ένωση Κεφαλαιογορών. Δεν είναι ένα προς ένα. Έτσι καταλαβαίνετε τι λέω. Πώς ε, βλέπετε τη σχέση αυτών των δύο ενώσεων, γιατί η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών δεν ταυτίζονται, αλλά θα έχουν πολύ πολύ στενή και πρέπει να είναι και πάρα πολύ γερή η σχέση που θα ε, τη συνδέει. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Για το τελευταίο που είπατε τη σχέση, τη σύνδεση. Η Ένωση της Κεφαλαγοράς είναι για το 28 όπως ξέρετε. Είναι για 28 χώρες. Και είναι ένα κλασικό πρόγραμμα ενιαίας αγοράς. Η Τραπεζική Ένωση έλυνε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που νομίζω έχει επιτυχώς επιλύσει ενώ η Ένωση της Κεφαλαγοράς αφορά ένα μια διαφορετικό πρόβλημα η Τραπεζική Ένωση υποστηρίζει, συμπληρώνει την άλλη αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αν και η Ένωση της Κεφαλαίου Αγοράς είναι πιο ευρία, έχει και τραπεζική, στοιχεία τραπεζικής ένωσης. Αλλά πάντως μια ενιαία αγορά κεφαλαίων και για τις 28 χώρες πρέπει να ωφελεί όλους και να συμμερίζονται όλοι τη λειτουργία του, να συμμετέχουν για την πτώχευση και τη φορολόγηση ή την αφαιρεγκαιότητα μάλλον. Θα επανέλθω και γι' αυτό με πιο συγκεκριμένες προτάσεις ε, για συγκεκριμένους τομείς. Ως επενδυτής βέβαια αν αντιμετωπίζετε πολύ διαφορετικούς νόμους για την πτώχευση σε κάθε χώρα, ε, αυτό εμποδίζει φυσικά τις επενδύσεις ε, ανεξαρτήτως χώρας. Η αρμόδια επίτροπος θα το επεξεργαστεί και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. κυρία Γιούροβα. Έχω συζητήσει με εκπροσώπους του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, χθες ναι. μάλιστα, και είδα ότι στα πλαίσια της Πράσινης Βίβλου θα επανέλθω για το θέμα, την λιανική πλευρά του θέματος για να τα ξαναδούμε αυτά και να διασφαλίσουμε ότι μερικά από τα μέτρα που έχουμε ήδη λάβει θα έχουν χορηγήσει περισσότερη προστασία, περισσότερα δικαιώματα στους καταναλωτές και να δούμε και τι θα λείπει. Στο με Παύλος Ζάνμπα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπόρεσα να ακούσω την παρέμβασή σας στην αρχή και θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και σε ό,τι φορά τη δική μου έκθεση. Σας συγχαίρω και για την πράσινη βίβλο. Είναι ένα καλό έγγραφο και καλό σημείο αφετηρίας. Μακάρι να γίνει και πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό, άμποτε. Σήμερα το πρωί Ήμουν στην πόλη μου στην Παμπλώνα και συμμετείχα σε μια εκδήλωση των σημαντικότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, της Ισπανίας και εξέφρασαν και πάλι την δυσφορία τους γιατί ε, αντιμετωπίζουν θέμα, δεν είναι αποκλειστικά της Ισπανίας αλλά είναι των νότιων χωρών που ε, είναι η έλλειψη πιστώσεων και εξαρτάται η επιβίωσή τους για πολλές και δεν τους εμποδίζει να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Συμφωνώ για όλα όσα είπατε για την ε, Ένωση Κεφαλαιογορών. Θα μπορούσατε να μου πείτε πώς θα εξηγήσω όμως σε ένα μικρομεσαίο, σε έναν εργαζόμενο εταιρεία πώς αυτή η Ένωση Κεφαλαιογορών θα τον βοηθήσει. Όταν του λέει όχι μια τράπεζα, να ξέρει ότι έχει άλλες εναλλακτικές. Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά που μας λέτε, έχετε όλη μου την υποστήριξη εγώ πείτε ότι είμαι μικρό επιχειρηματίας. Πώς θα πάω να βρω λεφτά όταν δεν μου δίνει η τράπεζα. Πώς ας πούμε κάποιο από την Γερμανία μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση σε έναν Ιταλό ή Ισπανό μικρό επιχειρηματία. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Σε λίγες εβδομάδες είμαι και στην Ισπανία και θα παρουσιάσω εκεί αυτό το εγχείρημα και ελπίζω να συναντήσω και εκπροσώπους μικρομεσαίων. Και με χαρά να ε, έχω μαζί τους ε, συζήτηση. Το πρώτο που θα σας έλεγα, που είμαι βέβαιος ότι το είπατε κι εσείς, είναι να τους ενθαρρύνω στη διαβούλευση να μας δώσουν όποιες πρακτικές ιδέες μπορεί να έχουν και προτάσεις, να συμμετέχουν στη διαβόλευση για να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις δικές τους ανάγκες. Η δική μου απάντηση είναι, στο βαθμό που μπορώ να βοηθήσω, ότι οι διάφορες εταιρείε στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους και της εξέλιξης έχουν διαφορετικές ανάγκες. Και σήμερα στα διάφορα κράτη-μέλη έχουμε οικονομική ανάκαμψη, υπάρχει το εκάστοτε σύστημα χρηματοοικονομικό που είναι σε διαφορετικά στάδια κάθε φορά. Υπάρχουν χώρες με ισχυρές τράπεζες και μικρομεσαίες πολύ συνδεδεμένες με τις τράπεζές τους και λειτουργούν καλά και πολύ καλά. Παρόλο που θα έλεγα ότι σε ορισμένες από τις χώρες αυτές που νομίζουν ότι λειτουργεί καλά, βλέπω ακόμα εκπροσώπους των μικρομεσαίων που μου λένε δεν μπορώ να βρω χρηματοδότηση, δεν μου δίνει δάνειο η τράπεζα. Πού μπορώ να βρω παρακαλώ άλλη εναλλακτική πηγή. Ε, στις αγορές, η, ο κεφάλαιο κινδύνου, οι ιδιωτικές επενδύσεις. Όταν είσαι μικρή επιχείρηση, και εγώ έχω τελές μικρός επιχειρηματίας στην αρχή, πήγα στην τράπεζα και τα βρήκα μπαστούνια και τελικά ανακάλυψα ότι υπάρχει και ιδιωτική επένδυση ε, με ε, τέτοια χρηματοδότηση σε μετοχές. Ε, η αγορά μπορεί να γίνει με διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, με τη δυνατότητα επιλογής ε, ε, των ανθρώπων ε, να, να μπορούμε και εμείς να αναπτύξουμε την αγορά. χρηματαγορές και άλλοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συμφέρον να χρηματοδοτούν και να ενημερώνονται. Είναι και θέμα πολιτισμικό καμιά φορά, κουλτούρας, νοοτροπίας. Εγώ όπως κι εσείς ε, πιστεύω ότι η κατάσταση πιέζει και είναι και επίγουσα, αλλά ορισμένα από αυτά έχουν να κάνουν με μια κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί χρόνια, χρόνια ολόκληρα. Και αυτό δεν αλλάζει ε, με νομοθεσία, με διατάγματα. Τώρα θα πας να δανειστείς από ιδιώτη, από κάποιον της κοινωνίας. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση για να αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει και η νοοτροπία. Ευχαριστώ. Thank you. Last speaker, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ Επίτροπε. Μια διαφορετική προσέγγιση έχω εγώ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για μια νομοθεσία ή κανονισμός που θα πρέπει να αντιστοιχεί στα προβλήματα της Ένωσης, να έχουμε οικονομική ανάκαμψη και απασχόληση. Αλλά ουσιαστικά αυτό λαμβάνει ως προϋπόθεση ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας λειτουργεί ανέκαθε λειτουργούσε υπέρ των επιχειρήσεων, υπέρ των καταναλωτών, υπέρ των πολιτών. Ουσιαστικά δεν θα πρέπει ο χρηματοπιστωτικό τομέας να λειτουργεί για να εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Βλέπουμε ότι στον χρηματοπιστωτικό τομέα υπάρχει ακόμα υπάρχουν ακόμα διαδικασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ πολύπλοκες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν δύναται αυτή τη στιγμή ο πολίτης να εμπιστευθεί το το χρηματοπιστωτικό τομέα. Εσείς ε, τι ρόλο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να δραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ανακάμψει η εμπιστοσύνη των πολιτών στο χρηματοπιστωτικό τομέα και τι ρόλο θα μπορούσε να δραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια πιο ήπια προσέγγιση που δεν θα είναι αναγκαστικά κανονισμοί, αλλά θα είναι για παράδειγμα κώδικες διοντολογίας, κώδικες συμπεριφοράς όσον αφορά για παράδειγμα τις τράπεζες. Προβλέπετε εσεί μια τέτοια προσέγγιση, τέτοια μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όσον αφορά τώρα την Ένωση Κεφαλαγορών, μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να διαχειριστούν περισσότερες πληροφορίες και μια πιο ευρύτερη ενημέρωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να δανειοδοτούνται και από άλλους φορείς, όχι μόνο από τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες κατέχουν τις περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απάντηση. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες αξίες, συγκεκριμένες αρχές, πρότυπα. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να τον σε θέση να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο του, να χρηματοδοτεί πραγματικά την ε, γενικότερη οικονομία και θα ήθελα πραγματικά να μπορούσα να πιέσω το χρηματοπιστωτικό τομέα να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι υγιής η φυστάμενη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, διότι βλέπουμε ακόμα ότι ε, πολλές φορές ε, ορισμένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν λειτουργούν θετικά για τις ίδιες τις χώρες ή για τους ίδιους επενδυτές τους. Πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι το βασικό μέρος της ευθύνης βρίσκεται στον ίδιο τον τομέα, τον χρηματοπιστωτικό. Πράγμα το οποίο σημαίνει θα πρέπει να αναλυφθούν, να υπάρχει κατάλληλη διοίκηση, ρύθμιση αν θέλετε του κανόνα αυτού θα μπορούσαμε εμείς εξωτερικά να επιβάλλουμε κάποιους κανόνες προκειμένου να έχουμε περισσότερη διαφάνεια, π.χ. στις αναφορές κτλ. Αλλά εν τέλει τελικά θα πρέπει οι αξίες αυτές να προκύψουν από τους ίδιους τους εργαζόμενους στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Δεν μπορεί η προσέγγιση μας να είναι μόνο ρυθμιστική, γιατί το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι ενδεχομένω να περιπλέκουμε εμεί τα πράγματα οι επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού κομμέα θα προσλαμβάνουν όλο και περισσότερους δικηγόρους για να δούνε πώς μπορούν να αποκριθούν στις δικές μας επαχθείς ρυθμίσεις, αλλά τα πράγματα δεν πρόκειται να λειτουργήσουν ποτέ θετικά κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει από τον ίδιο το χρηματοπιστωτικό τομέα να προκύψουν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες. Και ο ίδιος ο χρηματοπιστωτικός τομέας γνωρίζει ότι αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές προκλήσεις. Όσον αφορά τώρα τις ενημερώσεις πιστοτικής φύσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σίγουρα πληροφορίες αυτές είναι πολύ σημαντικές και πολύ σημαντικό το ζήτημα το οποίο θίγεται. Όντως, επί του παρόντος είναι οι τράπεζες αυτές οι μόνες που έχουν τις πληροφορίες αυτές, που θα επέτρεπαν δηλαδή στις μικρομισές επιχειρήσεις να συνάψουν δάνεια στο εμπράστη λοιπόν βίβλο μας προσπαθούμε να δούμε αν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο σύστημα με συγκρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην επιβάλλουμε δηλαδή εκ των άνω ένα σύστημα το οποίο θα είναι ιδιαίτερα επαχθές και πολύπλοκο. Γιατί ενδεχομένω να έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν θέλουν βασικά να επενδύσουν, που δεν θέλουν να συνάψουν δάνεια και θα βρεθούν και αυτές μπλεγμένες σε ένα πολύ επαχθές ε, άκαμπτο σύστημα. Πάντως, αν εσείς έχετε συγκεκριμένες ιδέες, να εμπνέεστε περισσότερο από την πραγματικότητα της χώρας σας, την Ολλανδία, είμαι στη θέση σας για να ακούσω τις ιδέες σας αυτές. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Επίτροπο Τζόναθαν Χιλ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα. Θα ήθελα να τονίσω ότι ε, και εμείς προσβλέπουμε στην πολύ θετική συνεργασία που έχουμε και να βάλουμε στο κέντρο ή δυνατόν τον ίδιο τον πολίτη, τον πολίτη δηλαδή στο κέντρο των χρηματοπιστωτικών αυτών υπηρεσιών να σε ευχαριστήσω και για την υποστήριξη που μας έχετε δείξει όσον αφορά διάφορους νομοθετικούς φακέλους. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ ειλικρινά. Colleagues, may I ask you... Συνάδελφοι, μήπως να καθόσασταν σιγά σιγά για να πάμε στις ψηφοφορίες μας. I ask colleague to... Παρακαλώ τους συναδέλφους να έχουν τις κάρτες τους, τα μηχανήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν έλεγχο πρώτα. Λοιπόν, κάρτες για να κάνουμε έναν έλεγχο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 one additional vote. Έχουν έναν υπεράριθμο. Okay, yes, you are fine. So it's fine. Okay, we close the vote. Πέρας. Τελος. So ECR also one. Και η ECR ψηφίζει ένας παραπάνω. Λούκε, also we have to count. Κύριε Λούκε. Α, δεν έχετε κάρτα, σας μετράμε λοιπόν χωριστά. Α, πάμε. Ρενάτε Σόρο, υποβολή εκθέσεων και διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων. Είναι σχέδιο νομοθετικής πρότασης. Τροπολογία υπαριθμών 118. Ψηφί ΠΕΡ. Κατά αποχές απορρίψετε. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 και 21 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική α πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής αρχίζει τώρα. Yeah, you can yeah. Two against more. Two against more, yes. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 141 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 141. Αρχίζει ψηφοφορία. One EPP Περσέβει ένας από το ΕΛΚ. Still one EPP too many. Ακόμα. Ακόμα. Ας βγάλει κάποιος το ΕΛΚ την κάρτα του. Ευχαριστώ, Μπορχαρτ. Πέρας. Και πάλι... Ε, ε, συν δύο κατά, γιατί είναι δύο συνάδελφοι χωρίς κάρτα. Ωραία. Λοιπόν, 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για την 150. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ακόμα από το ΕΛΚΑ ένας παραπάνω ψηφίζει. Φέρες. Απορρίπτεται. Α, όχι, όχι, έχουμε συν δύο υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος. Άρα, θα πάμε τώρα στην 32 της η υπέρ, του εισηγητή συγγνώμη, κατά αποχέ εγκρίνεται, 33 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, είναι συμβατή με την 154 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 155 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος γιατί είναι 155 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Τι θα γίνει με το ΕΛΚ ε, που ψηφίζει ένας παραπάνω κατά αυτό. Πέρας. Συν υπέρ ή κατά. Συν 2 υπέρ, παρόλα αυτά απερίφθη. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά Νομίζω ότι θέλει έλεγχο. Μάλλον έχει απορριφθεί, αλλά στο λέξω. Δηλαδή εγκριθεί διορθώνει ο Πρόεδρος. Συν δύο στους υπέρ, το ΕΛΚ συνεχίζει να έχει έναν υπεράριθμο. Πέρας. Εγκρίνεται. This was 158, correct? 35. 35 πέ, Κατά αποχές απορρίπτεται. 36. Τι θέλετε για την 35, έλεγχο. Νομίζω ότι έκανα λάθος. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος γιατί 35. Αρχίζει τώρα. Mm -hmm. Πέρασε. Απορρίψετε. 36 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας. Αποχές. Απορρίπτεται. 159 πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ κατά απόχες έλεγχος γιατί είναι 167. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. One EPP too many. Το ΕΛΚ εξακολουθεί να έχει έναν υπεράριθμο. Πέρας. Plus two in favor. Συν δύο υπέρ. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ. Κατά. Με την ίδια πλειοψηφία κανονικά. Ας το ελέγξουμε όμως αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Κανονικά πρέπει να έχει εγκριθεί νομίζω. Αν δεν απατώμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές με την ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε καλά. Αρχίζει η ψηφοφορία. 170. No, because they are these again. See. So two more against. So it's rejected. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H με προφορική τροπολογία. Πρώτα θα ψηφίσουμε την προφορική, ψήφι υπέρ της προφορικής τροπολογίας, κατά. Νομίζω απορρίπτεται. Έλεγχος για την προφορική αρχίζει τώρα. Το ΕΛΚ εξακολουθεί να έχει έναν βουλευτή πέρα. Ευχαριστώ, Μπορχάρτ. Πέρα. Απορρίπτεται. Και τώρα τη συμβαστική χωρίς προφορικές τροπολογίες είπε Κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 117 αρχής ψηφοφορία. το ΕΛΚ να βγάλει μια κάρτα. Πέρας. Additional favor, I suppose. Mr. Luke. Κύριε Λούκε, είστε υπέρ, εγκρίνεται λοιπόν, είναι συν δύο τα υπέρ. Συμβαστική ΑΙ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 203 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. συμβαστική J με δύο προφορικές τροπολογίες, θα ψηφίσουμε πρώτα την πρώτη της ΓΚΟΕ, ψήφι υπέρ της πρώτης, κατά, αποχές, απορρίπτεται η πρώτη προφορική, δεύτερη προφορική τροπολογία των πρασίνων, υπέρ, κατά, νομίζω απερίφθηκε αυτό, αλλά ας το ελέγξουμε, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ένας απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το συμβασμό J χωρίς της ε, όπως ε, τροποποιήθηκε σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία περίθμων 205. Ψηφίπε κατά αποχές απορρίπτεται. 206. Είναι ταυτόσημη, εντάξει δεν την ψηφίζουμε. 57 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται 81 και 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά νομίζω ότι έχει εγκριθεί η ΣΥΑΡ και άλλοι είστε υπέρ εγκρίνεται 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά έλεγχος για την 83 άρχεται η ψηφοφορία I think you rejected e too many. Πάλι μία επιπλέον ψήφος από το ΕΛΚΑ, πέρας, απορρίπτεται. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 222 άρχιτη ψηφοφορία. Πάλι επιπλέον μία ψήφος από το ΕΛΚ. Εξακολουθεί είναι υπεράρθμα το ΕΛΚ. Πέρας. Εγκρίνεται. 223 ταυτόσιμη υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 225 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 226 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 227 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 228 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί 85, τροπολογία 86 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 230, 231 μάλλον υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 232 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 233 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 234 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 235 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 236 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 238 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 239 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 242 υπέρ κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Το ECR και η άλλη είναι κατά έτσι δεν είναι, άρα απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Όχι. Περνάμε στη συμβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ, κατά, αποχές, η Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 94 νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο το ελέγξουμε άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Όχι, εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 95. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο 98 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 98, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται, έχουμε ψηφία. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά Ψηφίζετε κατά, μάλιστα. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση και η τροπολογία 6, άρχεται ψηφοφορία. Πάλι υπεράριθμο του ΕΛΚΑ, πέρας και εγκρίνεται, εγκρίνεται σαφώς. Τροπολογία 7, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103, υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 103 άρτη ψηφοφορία πάλι υπεράριθμο του ΕΛΚ μια επιπλέον ψήφος πέρας δύο επιπλέον υπέρ, άρα εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 105, υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 111 Πάλι μια επιπλέον ψήφο από το ΕΛΚΑ. Πέρα. Απορρίπτεται. 113. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 116. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, άρτη ψηφοφορία. Πάλι μια επιπλέον ψήφος από το ΕΛΚ. Εξακολουθεί το ΕΛΚ είναι περάριθμο κατά μία ψήφο. Πέρας. 47 υπέρ, 2 κατά και 6 αποχές. 49 μάλλον, αν συμψηφίσουμε και τις δύο επιπλέον ψήφους. Τώρα Αρχίζουμε πάλι νομαστική ψηφοφορία για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, άρθρο ψηφοφορία. Πέρας. Το ίδιο αποτέλεσμα. Και ψηφίσουμε για την απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73 του κανονισμού. Απόλυτη πλειοψηφία χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Άρτη ψηφοφορία. το ψήφι υπέρ, συν 2, άρα 50 υπέρ, 5 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή μας. Και αποφασίσαμε επίση ότι θα ξεκινήσουμε άμεσα διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη έκθεση, γνωμοδότηση για Πεκόφολτα σχέδιο γνωμοδότηση με θέμα συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσει για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Είστε έτοιμοι? Ωραία. Συμβαστική τροπολογία α σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά Ελέγχουμε για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής α, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 26 συν 2 υπέρ, 28 υπέρ, άρα απορρίπτεται. Σωστά, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα της συμβαστικής α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία B σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής Β, άρθρη ψηφοφορία. Πάλι μια επιπλέον ψήφος από το ΕΛΚ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά για τροπολογία 26. One Υπεράριθμο πάλι το ΕΛΚ κατά μία ψήφο. Δεν καταλαβαίνω γιατί επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα, τέλο πάντων. Εγκρίνεται πάντως η τροπολογία. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 23. άρθρη ψηφοφορία. rapporteur was in Yes, but the rapporteur changed his mind. Okay. Yes. Vote is closed. Πέρας. Δύο ψηφία επιπλέον υπέρ και απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία C. Χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της C ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά Ελεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 31 αυτή ψηφοφορία. Υπεράριθμο πάλι του ΑΕΛ κατά μία ψήφο. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 39. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. ισοψηφία, αλλά προσθέτουμε και τις δύο επιπλέον ψήφους. Πρεμόζεστε κατά λου και κατά απορρίπτεται. Περνάμε στη βασική τροπολογία D, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Α, με προφορική τροπολογία, να ψηφίσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την προφορική τροπολογία, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Δύο επιπλέον ψήφοι κατάρα απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 51 Έχουμε και δύο επιπλέον ψήφους κατά, αλλά παρόλα αυτά εγκρίνεται η τροπολογία. Συμβαστική τροπολογία η υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 60, υπέρ, κατά. Α, ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 60, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία F, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 68, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 68 άρτη ψηφοφορία. Πάλι μια επιπλέον ψήφο του ΕΛΚ, πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 77, υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 77, άρτη ψηφοφορία. εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση και για την 78. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία H, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 88, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 88 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία I υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 Με συγχωρείτε, έτοιμα ξεχωριστής ψηφοφορίας για τροπολογία 107, υπέρ της 107. Προβλεπόταν στο τμήμα του συμβιβασμού I. Ψηφίσουμε ξεχωριστά την 107, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 109, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 109, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Προσθέτουμε μία ακόμα ψήφο και εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 110 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έχουμε δύο επιπλέον υπέρψηφου, σε κάθε περίπτωση πάντω απορρίπτεται. Λόγω ισοψηφία. Η 111 έχει αποσυρθεί, περνάμε στην 112. Υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 112, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 118. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία J, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 128. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 128 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Έχουμε δύο επιπλέον ψήφους που είναι κατά, άρα απορρίπτεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 141, 2 και 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται 149 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για τα 149 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση και για την 150. Πέρας. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μάλλον ηλεκτρονική επαλήθευση για την 153 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία, μάλλον, 160 υπέρ, κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 160. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Όχι. Όχι. Ναι, ναι είναι γνωμοδότηση βέβαια, γνωμοδότηση. Ναι, ναι. Υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά όχι ονομαστική. Μάλιστα. Πέρας. τέσσερις ψήφοι υπέρ, 13 κατά και 9 αποχές. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Πρωτού κλείσει συνεδρίαση θα είμαι πολύ σύντομος όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμής προβλέπεται ο τρίλογος στις 26 Μαρτίου, μάλλον να έχει ακυρωθεί, διότι ο Αντώνιο Ταγιάννη είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει, για τις 16, θα γίνει στις 16 Απριλίου η περίληψη των συστάσεων που έγιναν σε συνεδρίαση των συντονιστών της 10ης Μαρτίου του 2015 μετά από την έκθεση Μάιστατ όσον αφορά τις προδιαγραφές υποβολής εκθέσεων χρηματοοικονομικών. Οι συντονιστές λοιπόν αποφάσισαν να διορίσουν μια μόνιμη ομάδα εισηγητών και σκιωδών εισηγητών η οποία θα λειτουργεί εκ περιτροπής προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να, να παρακολουθεί καλύτερα τη δουλειά που γίνεται για το IFRS. Scrutiny Lots όσον αφορά τον Απρίλιο. Θα ασχοληθούμε πρώτα με την γνωμοδότηση και την έκθεση της EBA για την ε, προσαρμογές όσον αφορά την αξιολόγηση πιστώσεων Επίσης πάλι η δημόσια διαβούλευση της CBA όσον αφορά τις κατευθυντήρες γραμμές, το σχέδιο κατευθυντήρων γραμμών για τις σωστές πολιτικές ε, αποζημίωσης στα πλαίσια της CDR4 και διαβούλευση όσον αφορά τις τεχνικές προταγραφές για τα κριτήρια καθορισμού των ελάχιστων απαιτήσεων για τα Own Fund Eligible Liabilities. θα γίνει παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια της δικής μας της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2015 προκειμένου να αναφερθούμε στην έναρξη της πλατφόρμας επίπεδου 2 όσον αφορά τους τίτλους, τα securities. Επίσης θα έχουμε μία έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας όσον αφορά τον κανονισμό χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και πώς μπορεί ο κανονισμός αυτός να οδηγήσει σε ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο για τις κεφαλαϊκές αγορές και την Ένωση Κεφαλαϊκών Αγορών. Επίσης, οι συντονιστές αποφάσισαν να συντάξουν προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαγορών. Όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, οι συντονιστές αποφάσισαν να εγκρίνουν προφορική ερώτηση προς την, προφορική, ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις γενικότερες κατευθυντήρες γραμμές που θα ακολουθήσει όσον αφορά κυρίως το ζήτημα της απασχόλησης προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητες ημερομηνίε για να γίνει οικονομικός διάλογος στις 15-16 Ιουνίου ενδεχομένως με τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, να αποσταλεί επίσης επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας για να γίνει οικονομικός διάλογος το πρώτο ήμιση του 2015, να συμφωνήσουν επίση με την προτινόμενη ημερομηνία της 5ης Μαΐου για να γίνει δημόσια ακρόαση της ΑΦΚΟ όσον αφορά τους ε, νέους κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης και τη θεσμική τους πτυχή. Δεν θα συνταχθεί έκθεση όσον αφορά τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και θα γίνει ένας στατιστικός διάλογος με την Γενική Διεύθυνση Eurostat. Τέλος. Οι συντονιστές ε, αποφάσισαν να ζητήσουν μια άδεια για να αυξηθεί ο αριθμός των μελών, είναι 10 τα μέλη αυτά τα οποία θα πάνε στην Ισπανία ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει... Μα όχι, έχουμε και την ακρόαση, έτσι δεν είναι. Θα γίνει από κοινού με την Επιτροπή Τάξα. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 30 Μαρτίου, 30 Μαρτίου θα έχουμε κοινή ακρόαση, παρουσία του Επιτρόπου Μοσκοβισή και θα ζητήσουμε ζητήματα φορολογικά. Και θα είναι παρόντες και συνάδελφοι από την Επιτροπή ΤΑΞ, την Νέα Ειδική Επιτροπή ΤΑΞ. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο πρόταση όσον αφορά τον τομέα τη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα έχουμε και μία συνεδρίαση της Επιτροπής μας ΕΚΟΝ την 3η 31 Μαρτίου το πρωί και το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεδρίαση. Yeah. Okay.